τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Down και κάνει ό,τι του αρμόζει για να μπορέσει να διατηρήσει την πολυμορφία στην Ένωση. Τώρα στην ε, ψηφοφορία. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την ε, απλοποιημένη διαδικασία της έκθεσης του κυρίου Σάμπανοτς σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Την θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Η πρόταση εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Σάμπανοτς. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου ε, Μπροκ σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ασία τη θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναρξη της ψηφοφορίας. Τέλος της ψηφοφορίας. Η έκθεση εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπρόκ. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ρέιντσελ σχετικά με τις ανησυχίες του Ιρλανδικού λαού σε ό,τι αφορά στη συνθήκη της Λισαβόνας, στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με ονομαστική κλίση έναρξης ψηφοφορίας παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Ρέιντζελ δεύτερη έκθεση του κυρίου Ρέιντζελ σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τις ανησυχίες του Ιρλανδικού λαού σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τη θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση έναρξη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια και πάλι στον κύριο Ρέιντζελ. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της ε, έκθεσης του κυρίου Τεσέιρα σχετικά με το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Τεσέρα. Και περνάμε στην ε, έκθεση του κυρίου Χάουιτ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Θα εξετάσουμε την ε, πρόταση ψηφίσματος και πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Έναρξη, παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 8 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά θα ήθελα να κάνουμε ένα έλεγχο για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 8 ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ έναρξη της ψηφοφορίας τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται Περνάμε στην τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ παρακαλώ. κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Περνάμε στην παράγραφο 41 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα παρακαλώ της παραγράφου 41 ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Περνάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε στην παράγραφο 60 κατά τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τροπολογία 4 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 4 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία αριθμός 5 υπέρ παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 93 κατά τμήματα και με ονομαστική κλίση. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. περνάμε στην παράγραφο 99 κατά τμήματα. πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 101 κατά τμήματα και με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναρξη της ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται επίση. Μετά την παράγραφο 101 θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σιλβέστρη που έχει να παρουσιάσει μια προφορική τροπολογία. Ο συνάδελφος κύριος Σιλβέστρης παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, μετά από την παράγραφο 101 θα ήθελα να προσθέσουμε μία παράγραφο. Υποστηρίζει ότι μεταξύ των δικαιωμάτων των γυναικών ε, ε, ε, εντάσσεται και το δικαίωμα της μητρότητας και το δικαίωμα δια... και απαγορεύεται να γίνεται διακοπή της μητρότητας όταν αυτή επιβάλλεται από ε, κοινωνικο-οικονομικούς λόγους. Πρέπει επίσης να προστατευτούν και τα δικαιώματα των νεογεννήτων. Ναι. ναι, είναι καθαρό ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των 40 βουλευτών, οπότε απορρίπτεται η προφορική τροπολογία του κυρίου Σιλβέστρη. Περνάμε. Ναι, κύριε Σιλβέστρη. Ήθελα, σεβόμενος φυσικά την Ολομέλεια, να θυμίσω ότι και αυτοί που σηκώθηκαν κάποτε υπήρξαν έμβρια. Προχωρούμε. Προχωρούμε. Δεν ανοίγουμε τη συζήτηση. Προφορική τροπολογία απορρίφθηκε και προχωρούμε στην ψηφοφορία. Επικεφαλίδα 18. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Λοιπόν, τροπολογία 6 ηλεκτρονικός ένελχος. Έναρξη της ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται θέτω τώρα σε ψηφοφορία την επικεφαλίδα 18 κατά τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές θα ήθελα να το ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της επικεφαλίδας 18 ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ παρακαλώ έχετε το λόγο Κυρία Ρης, έχετε το λόγο. Έχετε ζητήσει το λόγο. Presidente, mi scusi, non posso... Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί δεν λειτουργούν τα ακουστικά μου. Μπορείτε να μου στείλετε... Ε, λειτουργούν τα ακουστικά. Ε, λοιπόν, δεύτερο τμήμα της παραγράφου 18, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 102. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 103. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 104. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος... We voted for both parts. Ε, παράγραφος 104, δεύτερο τμήμα. Με συγχωρείτε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 105, με χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 106 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της παραγράφου 106 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 106 με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ έναρξη λήξη ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας, γιατί θα καθυστερήσουμε με τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Κατά. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. να ελέγξουμε αλλά είναι πιο απλό να σηκώνετε τα χέρια. Τροπολογία 8. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 112. Ο κύριος Ταβάρες έχει να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 112. Κύριε Ταβάρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε- Πρόκειται για μια προσθήκη, λέει ο κ. Σταβάρης, στην παράγραφο 112 και θα την διαβάσω στα αγγλικά. Θεωρούμε θετικό το ότι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών για τους ηθαγενείς πληθυσμούς και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των ε, δράσεων αυτών και σε επίπεδο επιμελητίας και σε επίπεδο τεκμηρίωσης και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να υποστηρίζει τη δραστηριότητα αυτή. Την προφορική τροπολογία που μας παρουσίασε ο κύριος Ταβάρες δεν υπάρχει αντίρρηση. Οπότε ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία του κυρίου Ταβάρες. και είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ παρακαλώ υπέρ κατά αποχές δεν σηκώνετε τα χέρια σας, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 9, παρακαλώ. Έναρξη. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 135 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 με ονομαστική κλίση έναρξη της ψηφοφορίας Δεν υπάρχει γερμανική μετάφραση, πληροφορούμαστε. έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα της μετάφρασης. Okay. Okay. Τροπολογία 11 με κλίση. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. και περνάμε στην ε, ψηφοφορία στο σύνολο της ε, πρότασης ψηφίσματος με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναρξη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Χάουιτ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διακόψουμε τώρα την ψηφοφορία για την πανηγυρική συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ.